Ο κύριο Βίλαντ. Συνεχίζουμε. επόμενε ψηφοφορίε. Πρόταση ψηφίσματος ε, για τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν. Έχουμε ε, σε δύο τμήματα το αρχικό υπέρ κατά το πρώτο τμήμα αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο ψήφισμα που αφορά την υπόθεση του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου Σίσελη. Ένα κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη υπόθεση απαγωγές και κακοποίηση γυναικών. Ένα ψήφισμα από έξι πολιτικές ομάδες, παράγραφος 6, σε έξι τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση αρχής τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το πέμπτο τμήμα της παραγράφου. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 6 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. Ε, τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Η τρία νομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται η ένα υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται δύο υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη έτσι ε, αρχίζει η ψηφοφορία είναι το αρχικό κείμενο ψηφίσατε όλοι Φέρας. εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ακολουθούν οι επόμενες ψηφοφορίες. Για... Ε, ξέρετε, την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Single Resolution Board, αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Για την πολιτική συνοχή το 2014-2020 είναι 7 πολιτικές ομάδες που έχουν ε, κάνει κοινό ψήφισμα. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. ψήφισμα για τι κατευθυντήριες γραμμές Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Πέντε πολιτικές ομάδες έχουν κάνει ένα ψήφισμα. Εννέα τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Α, θα χρειάζεται έλεγχο αυτό. Αρχίζει η ηλεκτρονική παρήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 10 τροπολογία ονομαστικά αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασα. Απορρίπτεται ή 11 ονομαστικά. Αρχίζει τώρα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11. Ο κύριος Τίλιτσκα ζήτησε το λόγο. Μικρόφωνο. Με μικρόφωνο παρακαλώ. μια προφορική τροπολογία, μια μικρή λεπτομέρεια στο όνομα της Άλντε και την στηρίζουμε τέσσερις πολιτικές ομάδες. Εκτιμούμε τη δουλειά με τους συναδέρφους ε, καθώς και την πρωτοβουλία του κυρίου Πίπερ, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στην παράγραφο 11, όπου σήμερα ως έχει προτείνουμε να μην ε, υιοθετηθεί η πρόταση από την Επιτροπή εκτός αν υπάρχει θετική γνωμοδότηση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε στην Επιτροπή μία δήλωση η οποία θα δώσει στο Συμβούλιο ε, ανεξάρτητων ε, επιπτώσεων αντικτύπου δεν μπορούμε να υποδείξουμε στην Επιτροπή τι θα πρέπει να κάνει. Προτείνω λοιπόν να λέμε ότι προτάσει δεν θα πρέπει να υιοθετούνται από την Επιτροπή εκτό εάν συνοδεύονται από γνωμοδότηση την οποία να έχει εγκρίνει το Συμβούλιο ε, ε, ε, Επιπτώσεων Αντικτύπου. Συγγνώμη, μελετών αντικτύπου. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 15, ονομαστική ψηφοφορία, ε, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17, το αρχικό κείμενο. Σε δύο μέρη το πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20 το αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στο ψήφισμα για την 25η επέτειο της, ε, συμφωνίας ε, των, ε, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ε, τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος ονομαστική ψηφοφορία και της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 4 αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία 11, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 19, αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21, το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Ε, το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 36. Αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Εκτιμώντας F σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχή της ψηφοφορίας. Νομίζω κρίνεται. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Λυπάμαι, πολλές αποχές δεν μπορώ να κρίνω. Αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονική, Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Q, το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρο ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματο όπω τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Φτάνουμε στο ψήφισμα για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Έχουμε ε, ένα ψήφισμα δύο πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 7. Ποιο είναι υπέρ, κατά Παρακαλώ άλλη μια φορά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. 67. Αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Αρχή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 60. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 61. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62. Αρχή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 65. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Αρχή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 82. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μάλλον ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 69 αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για το δεύτερο μέρος. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Αρχή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 13 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14 σε δύο μέρη το αρχικό κείμενο. Υπέρ, πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η κυρία Κέπχαρτ. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά στο κατάλογο ψηφοφορία μας έχει πάρει σφρίσει ένα λάθος. Θέλαμε να υπερψηφίσουμε και όχι να καταψηφίσουμε. Είμαστε υπέρ το να έχουν τα άτομα με αναπηρία τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ευχαριστώ κύριε Κέπχαρτ. 19 ονομαστικά ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή τώρα. Έρχεται η ψηφοφορία. Το ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Βοήθησε κυρία Γκέπαρτ αυτό που είπατε. Πολύ αποτελεσματικό. Εγκρίνεται. Ε, ε, Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές. Α, υπέρ ξανά. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε για την 20. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 63 τροπολογία υπέ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 κλίση Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ε, ψηφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφθεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος χρειάζεται εδώ. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία παριθμών 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ ψηφίζετε, δεν είναι σαφές. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό χρειάζεται έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονική για την τροπολογία 39. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 Θέλετε έλεγχο για τη 45 ορίστε αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 είπε, Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 48 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 είπε. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 50 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 51 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει ψηφοφορία τώρα για την τροπολογία 51. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Α, έτσι να παληθεύσουμε την 57 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισα τέλο. Πέρασα. Μα το είχα δει ότι είχε εγκριθεί. 58. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεν είσαι Υπέ. Κατά. Τώρα δεν βλέπω τίποτα όμως. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, χρειάζεται έλεγχο. Αρχίζει η ηλεκτρονική παρήθευση. Μια μεγάλη ομάδα δεν ψηφίζει, μάλλον η ίδια πλειοψηφία θα είναι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε έλεγχο για την 25 ορίστε αρχίζει η υπαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Γκρίνεται. Ε, κάποιοι δεν είδανε καλά. Λοιπόν, το σύνολο ονομαστικά ψηφίζουμε τώρα που τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Angenommen. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο τελευταίο ψήφισμα. Υποσυντισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παράγραφος 10. Τροπολογία 1. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Ε, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα για την τροπολογία αυτή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Η τροπολογία 4. Π. Κατά. Α, ζητώ συγγνώμη, είναι ονομαστική αυτή. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απέριφθη. Οι δύο υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά ψηφίζουμε τώρα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ αφήστε τις κάρτες σας στο μηχάνημα μέσα μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ich möchte alle sehr herzlich bitten, Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους θερμότατα den Saal zu verlassen, die gehen möchten und sich unter όλους όσοι αποχωρείτε και θέλετε να έχετε ιδιωτικές συνομιλίες, να το πράξετε ησύχω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να ακούσουν τις επεξηγήσεις ψήφου. Και αυτοί παρακαλούνται να καθίσουν ξανά γρήγορα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας και τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν διατεθεί. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι. Είμαστε στις επεξηγήσεις ψήφου.